Pan Przewodniczący! Good morning, ladies and gentlemen. Ο Πρόεδρος, καλημέρα σας λέει και σας ζητώ συγγνώμη για αυτή την καθυστέρηση. Είχαμε μια συζήτηση πάρα πολύ συναρπαστική και ενδιαφέρουσα με τον κύριο Μπαρόσο και με τον κύριο Λεβαντόφσκι αλλά και τους αρχηγούς των πολιτικών ομάδων. Επομένως, γι' αυτό και καθυστερήσαμε λίγα λεπτά. Όμως, αυτή η συζήτηση που η οποία τώρα πρόκειται να γίνει είναι πάρα πολύ σημαντική.